και στις προσπάθειες που θα γίνουν ε, στη συνάντηση που θα γίνει στο Μπουτάν. Ευχαριστώ. Πέρα στη συζήτηση και θα ψηφίσουμε αύριο στις 12.30. Το επόμενο σημείο στη μερίσια διάταξη είναι η, κυρία, ε, είναι η έκθεση της κυρίας Σίμερ για την ενίσχυση των ε, αναπτυσσομένων χωρών στο να αντιμετωπίσουν τις επιθετιστικές προκλήσεις και ανάγκες. Ο εισηγητής έχει το λόγο για τέσσερα λεπτά η ναι, κυρία Τσίμερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε, και κύριοι. Σε μια επίκληση που ξεκίνησε με πρωτοβουλία Αφρικανών συγγραφέων για το κέρας της Αφρικής λέει ότι χρειάζονται οι άνθρωποι του κέρατος της Αφρικής τη βοήθεια όλων των ανθρώπων γιατί έχουν δικαίωμα σύμφωνα και με το άρθρο 25 της ε, Παγκόσμια διαχείριση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, δικαίωμα στην τροφή. Μιλούμε για εκατομμύρια ανθρώπων. Στην Σομαλία και μόνο τους τελευταίους μήνες πέθαναν πάνω από 30.000 παιδιά νεότερα των 5 ετών και οι άνθρωποι που πεινούν ανά τον κόσμο φτάνουν τους πάνω από το 1 δισεκατομμύριο. Με την επεξεργασία της εκθέσεως που έχω καταθέσει, τα μέλη της Επιτροπής Αναπτύξεως για αυτήν μάλλον βασίστηκαν σε δύο βάσεις. Αφενός το ερώτημα, η Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνει αρκετά σοβαρά υπόψη της τις ευθύνες της για να διασφαλιστεί η διατροφή των ανθρώπων από τον κόσμο. Το ίδιο για το καθαρό νερό, για την ενέργεια. Και δεύτερο, η Ευρωπαϊκή Ένωση πώς θα εξασφαλίσει την απαραίτητη συνοχή στις πολιτικές της ώστε να υλοποιηθεί ο στόχος που προβλέπεται και στα άρθρα 7 και 208 της συνθήκης της Λισαβόνας. Έχοντας υπόψη τις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του περσινού χρόνου για την υποστήριξη από πλευράς χωρών μελών και για την ανθρωπιστική βοήθεια στον τομέα των επισητιστικών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει βάλει ορισμένες προϋποθέσεις, τις οποίες υποστηρίζουμε εμείς ως Επιτροπή Αναπτύξεως. Από την άλλη μεριά εκτιμούμε ότι σε πολλού τομεί οι προσανατολισμοί αυτοί δεν είναι επαρκείς. Για παράδειγμα, Πού βρίσκεται η απαραίτητη συνοχή μεταξύ όλων των πολιτικών, ιδίως για την διεθνή εμπορική πολιτική, για την αναδιάρθρωση της αγροτικής πολιτικής, εκεί όπου πρέπει να γίνουν απαραίτητες διορθώσεις. Ένα άλλο μεγάλο έλλειμμα είναι ότι ο αγώνας κατά της πείνας στον κόσμο δεν έχει λάβει αρκετά υψηλή προτεραιότητα στους διάφορους διεθνείς οργανισμούς, ούτε άλλωστε και στην πολιτική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η λοιμή οι καταστροφές πείνας δεν έρχονται από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι σαφές αυτό και από το περιεχόμενο της έκθεσής μας. Είναι σαφές επίσης ότι η αλλαγή του κλίματος, η κερδοσκοπία στα χρηματιστήρια, η τιτικότητα των τιμών, η αρπαγή των υγειών, όλα αυτά αποβαίνουν πρωτίστως σε βάρος των φτωχότερων από τους φτωχούς των προσφύγων, των απροστάτευτων γυναικών και παιδιών, των υπερηλίκων. Εμείς ρίξαμε το βάρος μας ιδίω σε τρία σημεία στην έκθεσή μα. Αφενό υποστηρίζουμε και θέλουμε να επεκταθεί αυτό ότι θα πρέπει να επιλεγεί μια προσέγγιση βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα για την εξασφάλιση της τροφή. Το ανθρώπινο δικαίωμα στην τροφή θα πρέπει να βρεθεί ως ύψιστη προτεραιότητα στην ατζέντα, την πολιτική ατζέντα και να προωθηθεί. Μια μικρή, σε μικρή κλίμακα γεωργία με χαρακτήρα διαρκή και βιώσιμο θα είναι η λύση. Χρειάζεται λοιπόν να γίνουν μαζικές ε, αυξήσεις των επενδύσεων στη γεωργία. Το ίδιο ισχύει και για συγκεκριμένα μέτρα για την εφαρμογή μέτρων ασφάλειας για την διατροφή και κατά της ανεξέλεγκτης αρπαγής γεών που είναι πολύ μεγαλύτερες οι διαστάσεις από ό,τι μέχρι τώρα θεωρούσαμε. Τα τελευταία νούμερα που έχουμε για την Ουγκάντα, για παράδειγμα, μιλούν για παραπάνω από 21.000 εκτοπισμένους από τις γέες τους, διότι οι γέες αυτές αγοράστηκαν από μεγάλες επιχειρήσεις. Τρίτο, και αυτό είναι το τρίτο μεγάλο θέμα, χρειαζόμαστε την απαραίτητη συνοχή στις πολιτικές, έτσι ώστε να μην γίνεται από τη μια μεριά πολιτική ανάπτυξη με διάθεση κονδυλίων στις χώρες αυτές, από την άλλη μεριά με άλλες εμπορικές πολιτικές να καταστρέφονται τα αποτελέσματα των πρώτων. Θα ζητήσω λοιπόν την υποστήριξή σας για την ε, έκθεσή μου στην αυριανή ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ. Η Πρόεδρος προχωρούμε στο σύστημα Catch the Eye με πρώτη την κυρία Αντωνέσκου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε ένα μεγάλο ανθρωπιστικό πρόβλημα γενικότερα και η επισητιστική, η επισητιστική ασφάλεια είναι ένα μεγάλος κίνδυνος και έλλειψη ασφάλειας στον ε, σημερινό κόσμο, ε, πίεση ε, στα υδάτινους πόρους, ένδια, λοιμός και χαιρετίζω την πρόταση να, να αποτελέσει το δικαίωμα στη διατροφή σε ένα ακρογωνίο της πολιτισμής μας. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μία πολύ ε, συνεχτική πολιτική σε όλα τα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης χρειαζόμαστε αναπτυξιακή πολιτική, ενεργειακή πολιτική, ερευνητικά προγράμματα και ε, εμπορική πολιτική να ε, συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια. Και θα πρέπει να υπάρχουν και διαφανείς ε, μηχανισμοί με συμμετοχή της ε, κοινωνίας των πολιτών και όλων των ενδιαφερμένων φορέων για να μπορέσουν να εφαρμοστούν σωστά όλες αυτές ε, οι πολιτικές. Ευχαριστώ. Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μετά θα μιλήσει ο Επίτροπος. Σε κάποιες περιοχές της Αφρικής υπάρχει αυτή η πρόκληση της έλλειψης διατροφής και ξέρουμε ότι υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι που πεθαίνουν από έλλειψη τροφής. Νομίζω ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση διαφορετικά θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε παγκοσμίω το πρόβλημα αυτό. Η συνειδητοποίηση του προβλήματος του εκ μέρους της παγκόσμιας κοινωνίας ήταν πάρα πολύ αργή. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ενισχύσουν σημαντικά την συμμετοχή του ώστε να μπορέσει η ανθρωπιστική βοήθεια να γίνει αναπτυξιακή βοήθεια, κυρίως να αναπτυχθεί η γεωργική ε, πολιτική, κυρίως η ανάπτυξη της υπαίθρου σε όλες τις χώρες αυτές. Επίσης, να υποστηρίξουν διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα με ευρεία συμμετοχή όλων όσων έχουν ανάγκη. Τέτοιου είδους προγράμματα εκπαιδευτικά θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα ε, αποτελεσματικό μέσων για να ξεφύγουμε από αυτή την ε, οδό χωρίς ε, διέξοδο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, η ασφάλεια των ειδών διατροφής στις αναπτυσσόμενες χώρες είναι θέμα ζωής ή θανάτου σε πολλές ε, χώρες σήμερα. Είναι λοιπόν ηθική υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επιλέξει τις κατάλληλες μεθόδους επιστημιστικής βοήθεια προς όλες τις χώρες και να βοηθήσει την αηφόρο παραγωγή ειδών διατροφής και όλες τις χώρες, δεδομένου ότι αυτό αποτελεί τη βάση της ανάπτυξης της ε, όλων των περιοχών και των λιγότερων ανεπτυγμένων χωρών. Τέτοιου είδους δραστηριότητες βεβαίως εξαρτώνται από την εξωτερική βοήθεια, κυρίως να λάβουμε υπόψη και τις ε, γυναίκες και όλου αυτούς που ζουν στι μικρά αγροκτήματα. Νομίζω ότι η κερδοσκοπία στην αγορά ε, πρώτων υλών, η αύξηση της τιμής των καυσίμων είναι καταστροφικές για τον τομέα αυτό και θα πρέπει κάτι να κάνει και η Επιτροπή να μπορέσει να, να διευθετήσει την ε, ε, κατάσταση αυτή. Ευχαριστώ κυρία Would... Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον εισηγητή για τη θαυμάσια έκθεση. Πιστεύω ότι η γεωργία είναι μία από τις πολιτικές όπου υπάρχει περιθώρια ανάπτυξης και κυρίως εκεί υπάρχουν και μεγάλες συγκρούσεις. Ε, δεν θρέφουμε τον κόσμο με έναν τρόπο που σχεδιάζουμε τώρα την αγροτική πολιτική. Και δεν νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε. Θα πρέπει η παραγωγή τροφίμων να γίνεται τοπικά, δεν θα πρέπει να ανταγωνιζόμαστε στις παγκόσμιες αγορές με την ευρωπαϊκή ε, αγροτική μας πολιτική. Δεν θα πρέπει να εστιάζουμε στον ανταγωνισμό. Αντίθετα, θα πρέπει να βοηθούμε τις αντισώμενες χώρες να τραφούν οι ίδιες. Τι κάνουμε όμως αυτή τη στιγμή. Η παραγωγή κρέατος μας κατά 72% ε, βασίζεται στην παραγωγή σόγιας, 20 ε, εκατομμύρια εκτάρια εξάγουμε, αλλά και εισάγουμε σόγια από 9 εκατομμύρια εκτάρια. Στην πραγματικότητα δεν τρέφουμε τον κόσμο, τον, τον σε λοιμό. Θα πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε την πολιτική μας, να κάνουμε μια εσωτερική ε, μεταρρύθμιση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η συζήτηση ενό στρατηγικού πλαισίου για να βοηθήσουμε τι αναπτυσσόμενε χώρε να αντιμετωπίσουν τι προκλήσει που έχουν σε θέματα επιστημιστική ασφάλεια είναι καλόδεχτη και βεβαίως όπως είπε και ο εισηγητής έχει μεγάλη σχέση με την συνεκτικότητα μεταξύ αυτής της πολιτικής και των πολιτικών των, ε, που κατά τομέα έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμπορική, ενεργειακή, γεωργική, εμπορική κτλ. Και σήμερα όντως υπάρχει μία μεγάλη ε, ασυνέπεια μεταξύ όλων αυτών των πολιτικών. Η ελεύθερο εμπόριο, η προώθηση ε, μοντέλων ε, εντατικής κατα... καλλιέργειας που καταστρέφουν τις οικογενειακές εκμετανεύσεις και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το γεγονός ότι δεν παράγονται σωστά τα ίδια τροφής, απειλεί την ε, επιστημιστική ανεξαρτησία και κυριαρχία των ε, μικρών χωρών. Όσο περισσότερο εξαρτώνται μικρές χώρες από βοήθεια και όσο περισσότερο εξαρτώνται από την προμήθεια από τις μεγάλες χώρες, τόσο περισσότερο θα συνεχίζουν να έχουν αυτές τις μεγάλες ανάγκες. Ευχαριστώ. Συζητάμε σήμερα μεταξύ των άλλων πώς θα διευκολύνουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες στο να αντιμετωπίσουν τα επισητιστικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Και από τη μια πλευρά και προσθέτοντας τα όσα είπαν οι συνάδελφοι χαράσουμε πολιτικές συζητάμε σήμερα την εξαιρετική έκθεση πράγματι της εισηγήτριας κυρία Ζήμερ και την ευχαριστούμε γι' αυτό ακούμε από την επιτροπή όλο το σχεδιασμό και τις πρωτοβουλίες. από την άλλη πλευρά όμως τον μάιο τον περασμένο μάιο στις 10 μαΐου η επιτροπή ανακοίνωνε ότι εξετάζει τη μείωση στο μισό και παραπάνω των χωρών που χαίρουν του συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων. αντιλαμβάνομαι πλήρως το νόημα αυτής της ανακοίνωσης και το έχω μελετήσει ρωτώ όμως την επιτροπή και θα ήθελα μια απάντηση πώς εναρμονίζονται αυτές οι ανακοινώσεις της επιτροπής με τη δέσμευσή μας για αύξηση της βοήθειας προς τις αναπτυσσόμενες χώρες. ευχαριστώ. Πάσκα. Ευχαριστώ. κύριε Πρόεδρε, γυναίκες και παιδιά είναι που υποφέρουν περισσότερο και οι μεγάλοι άνθρωποι. Αυτό είναι το σημαντικότερο συμπέρασμα από την έκθεση. Ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι πρέπει να παραμείνουν οι αρρώσιμες γέες στα χέρια των τόπιων πληθυσμών. Οι δεμοί οδηγούμαστε σε ανεξέλεγκτη μετανάστευση των προσώπων αυτών προς τα αστικά κέντρα. Οι κυβερνήσεις πουλώντας τις γέες στερούν από τον πληθυσμό τους τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν τα, την απαραίτητη, τα απαραίτητα Έχουμε λοιπόν ηθικό καθήκον να ζητήσουμε να αρχίσει διάλογος για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ την κυρία Τσίμερ για την έκθεσή της, καθώς και όλους τους ευρωβουλευτές για τις παρεμβάσεις τους για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Είμαι χαρούμενος που η κυρία Τσίμερ συμφωνεί με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την βοήθεια προς τις αναπτυσσόμενες χώρες να αντιμετωπίσουν τις ε, προκλήσεις της επιστικής ασφάλειας που δημοσιεύθηκε το Μάρτιο του 2010 και από τις προτεραιότητες που αναφέρει αυτό το πλαίσιο. Θα γνωρίζετε ότι η πρόσφατη δημόσια συζήτηση για το μέλλον της ε, αναπτυξιακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντόπισε ότι η γεωργία και η επιστημιστική ασφάλεια είναι οι βασικοί τομεί όπου θα πρέπει να ε, προωθήσουμε τη βιώσιμη και την πράσινη ανάπτυξη. Αυτή η επιστημιστική ασφάλεια είναι προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία είναι δεσμευμένη απόλυτα να υποστηρίξει του εταίρου τη στο να επιταχύνουν τι επενδύσει για να υπάρξει αυτή η ασφάλεια. Πιστεύουμε ότι υπάρχει πραγματικό δυναμικό για να αναζωογονήσουμε τι αναπτυσσόμενε χώρε, ούτω ώστε να γίνει πρόοδο για την υλοποίηση των στόχων της ε, χιλιετίας. Ε, το πρόβλημα είναι όλο και πιο ανησυχητικό, ε, οι προκλήσεις όλο και μεγαλύτερες. Η σημερινή κατάσταση στο κέρας Αφρικής δείχνει μια φρικτή εικόνα και μας δείχνει ότι είναι και η ώρα να δράσουμε από κοινού για να δώσουμε απαντήσεις και λύσεις και στην βραχυπρόθεσμη, στο βραχυπρόθεσμο πρόβλημα, αλλά να αντιμετωπίσουμε και πιο μακροπρόθεσμα το πρόβλημα. Θα πρέπει να έχουμε λοιπόν ε, να εξασφαλίσουμε την επιστηστική ασφάλεια με τον πιο βιώσιμο τρόπο για τους πιο ευάλους πληθυσμούς και να τους βοηθήσουμε να ε, δείξουν μεγαλύτερη αντοχή. Για μας είναι προτεραιότητα και θα εξακολουθήσει να είναι και κυρίως η γεωργία. Σε ό,τι αφορά τις ανησυχίες που αναφέρει το ψήφισμα για την ε, οικονομική κερδοσκοπία και την εξαιρετική αστάθεια των τιμών στα τρόφιμα, εμείς ε, εξετάζουμε το επίπεδο της κερδοσκοπίας και το επίπεδο και την αστάθεια των τιμών των τροφίμων. Ούτως ή άλλως θα πρέπει να υπάρχει και διαφάνεια στην αγορά και να την εθαρρύνουμε, ούτως ώστε να λειτουργούν καλύτερα οι αγορές και να μπορούμε να δρούμε καλύτερα και με πιο συντονισμένο τρόπο. Σας διαβεβαιώ ότι η Κομισιόν παρακολουθεί πολύ προσεκτικά την κατάσταση της αύξησης των τιμών των τροφίμων και τις επιπτώσεις που υπάρχουν στις ε, αναπτυσσόμενες και ευάλωτες οικονομίες και θα λάβει δράση η αναθεώρηση δύο σημαντικών νομοθετικών κειμένων, ε, ο κανονισμός για τις χρηματαγορές ε, και η οδηγία για τις ε, καταχρήσεις της αγορές είναι εν εξελίξη και οι προτάσεις της Κομισιόν θα γίνουν το φθινόπωρο. Τα μέτρα θα αφορούν την αύξηση της διαφάνειας και της ακαιρεότητας των χρηματαγορών θα αφορά και την αγορά των γεωργικών παραγόγων. Επίσης, η επιστημιστική βοήθεια θα πρέπει να δίδεται με τον πιο δυνατό τρόπο, ε, με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Έχουμε κάνει μια δήλωση προθέσεων για αυξημένη ε, συνεργασία με, τους, ε, με τις τρεις υπηρεσίες του ΟΗΕ που βρίσκονται στην Ρώμη. Σας διαβεβαιώνουμε ότι θα πρέπει να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα των ανθρώπων που μισθώνουν, που κατέχουν δηλαδή προσωρινά τη γη και δεν θα πρέπει αυτά να διακυβεύονται από μαζικές εξαγορές γεών. Επίσης, θα πρέπει να έχουμε τις κατάλληλες ε, πολιτικές για τη γη σε διεθνές επίπεδο. Πιστεύουμε ότι η βιώσιμη αλία και η ηχθειοκαλλιέργεια μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση του λοιμού και της κακής διατροφής. Και θα παραμείνουν προτεραιότητες της αναπτυξιακής συνεργασίας. Όλοι συμμεριζόμαστε αυτές τις απόψεις. Θα είμαστε παρόντες στην ε, ακρόαση που οργανώνει το Κοινοβούλιο για την επιστηστική ασφάλεια την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Κλείνει η συζήτηση. Θα ψηφίσουμε αύριο στις 12.30. Και τώρα περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης που είναι η έκθεση του κυρίου Καβαντά για το σύστημα των Ευρωπαϊκών Σχολείων Κύριε Καβαντά, έχετε το λόγο για τέσσερα